κοινοβούλιο χωρίς βουλευτές. Ε, καλή σας όρεξη κύριε Κέλλη και ε, στις υπηρεσίες και στους διερμηνείς. Ε, καλή σας όρεξη, διακόπτη τη συνεδρία.